ένα έτος πρακτικής εφαρμογής πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων πολιτών. Αξιολόγηση εμπειρών και, και αντιμετώπιση εμποδίων. Ωραιότατος τίτλος. Κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε αυτή την αξιολόγηση και να ξεπεράσετε και τα εμπόδια και να τα αντιμετωπίσετε. Αξιότιμοι βουλευτές, ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω εν συντομία όχι την πρώτη αποτίμηση αλλά τις πρώτες σκέψεις που έχουμε μετά την ε, θέσπιση της ε, πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι ε, πολύ προώρο να καταλήξουμε συμπεράσματα. Είναι καλή ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε και να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και επίσης να τροφοδοτήσουμε το μιλοντικό μας προβληματισμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δραστηριοποιήθηκαν και για τη θέσπιση και για την υλοποίηση του στόχου μας. Οι πρώτοι 12 μήνες ε, δεν δημιουργήσαν ε, τόσο μεγάλα εμπόδια. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για αυτό το εργαλείο συμμετοχική ε, δημοκρατία. Ευρέως ήταν θετική η εμπειρία και γίναμε μάρτυρε ενό φαινομένου που έχει προοπτική να αναδειχθεί σε ένα ισχυρό εργαλείο, ούτω ώστε να εμπλακούν άμεσα οι πολίτε σε εργασίες των θεσμικών οργάνων τη Ένωση. Η πρωτοβουλία των πολίτων μπορεί να είναι πηγή αισιοδοξία ε, θέλουν να ακούγεται η φωνή του και να εμπλέκονται οι πολίτε. Άρα χρειάζονται και τα πετούμενα μέσα για να το πετύχουν. Ε, και παρότι δεν μπορούμε να προδικάσουμε την έκβαση οποιασδήποτε πρωτοβουλία, θεωρούμε ότι αξίζει τον κόπο. 14 πρωτοβουλίε έχουν καταγραφεί προ στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλύπτουν το φάσμα, ΜΜΕ, ε, δημόσιε υπηρεσίε, παιδεία, δοκιμέ με ζώα, κλιματικέ αλλαγέ, όρια ταχύτητα και και ούτω καθεξής. Ε, και στη Δύο εκατομμύρια υπογραφές έχουν συλλεχθεί για αυτά τα θέματα. Πέραν αυτού φαίνεται ότι δραστηριοποιούνται διασυνοριακά ε, οι πολίτες ε, των κρατών μελών και τροφοδοτείται και ο δημόσιος διάλογος για τόσο σημαντικά ζητήματα και αυτό είναι και το ζητούμενο για μας. Φυσικά είχαμε και δυσκολίες, είχαν ε, προέκυψαν προβλήματα με τα ΜΜΕ, παραδείγματο χαρή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη εργάστηκαν πολύ σκληρότερα σε σχέση με τι αρχικέ προβλέψει, ώστε να είναι ταχύα και αποτελεσματική η εφαρμογή αυτή τη ε, πρωτοβουλία. Ε, το ίδιο ισχύει για όλου του εμπλεκόμενου φορεί. Θα ήθελα να τονίσω κάποια ζητήματα όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να αντιμετωπίσει τα εμπόδια και να διευκρινίσει κάποιε παρανοήσει που προέκυψαν. Όταν θεσπίστηκε η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία τον Απρίλιο του 2012, πριν από ένα χρόνο, ε, λίγανε με έναν τέτοιου είδους ε, δυσκολίες, ε, ούτως ώστε να έχουμε τους φορείς που θα μας βοηθήσουν με την επιστοποίηση της επιγραμμικής συλλογής ε, υπογραφών ε, και ως προσωρινή μεταβατική λύση προ, προ, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δωρεάν με τις υπηρεσίες στο Λουξεμβούργο να προσφέρει επιγραμμική συλλογή υπογραφών και για να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο αναλάβαμε τη δέσμευση επίσης ε, να ε, λάβουμε υπόψη την ε, συλλογή πέρα, μετά την εκπνοή της 12μηνης περίοδου, δηλαδή μετά το Δεκέμβριο του 2013. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα μέτρα είχαν σημαντικό αντίκτυπο ως προς το χρόνο και την ενέργεια που έπρεπε να επενδύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατέβαλε σημαντικότερες προσπάθειες για την κατάρτιση, την καθοδήγηση, καθόλου την διάρκεια της διαδικασίας και εκτεταμένα διαβουλεύτηκε με τα κράτη-μέλη, ώστε να συνυπολογιστούν και δικέ του ανησυχίε αντιμετωπίσαμε αυτές τις ανησυχίες και μπορούμε να αναμείνουμε τώρα ε, στο μέλλον ε, τεχνικός ε, και διοικητικός πώς να είναι καλύτερη η οργάνωση. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερεύει κατά πολύ τα προβλεφθέντα από την νομοθεσία με τρόπο ώστε να επιτύχει αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών. Μπορεί θα έλεγαν ότι αν ήταν λιγότερο αυστηρέ οι διατάξει του εκτελεστικού κανονισμού, θα ήταν ευχερέστερη η διαδικασία. Ενδέχεται να αληθεύει αυτό, αλλά πρόκειται για προσωπικά δεδομένα. Έχουμε την ασφάλεια, τι τεχνικέ προδιαγραφέ για να ε, διαφυλάσσουμε το απόρριτο για του υπογράφου, αλλά και η όλη διαδικασία συλλογή ε, υπογραφών ε, είναι δυσχερή διαδικασία. Τίποτα δεν είναι θέσφατο βεβαίω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαβουλεύονται για οποιαδήποτε απόφαση αναθεώρηση ούτω ώστε να βασιζόμαστε σε πραγματικά στοιχεία. Φυσικά ενδεχομένω ε, να χρειαστεί αυτή η αναθεώρηση, αλλά θέλουμε να παραμείνει αποκεντρωμένο σύστημα αυτό τη υποδοχή και συλλογή των υπογραφών ε, ή ε, να χρησιμοποιήσουμε ένα νέο κεντρικό σύστημα. Σε σχέση με το λογισμικό που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συλλογή των υπογραφών, ε, μα είπαν οι εμπλεκόμενοι ότι δεν βοηθάει αυτό το σύστημα. Ο αντιπρόεδρο Εύκοβη μα είπε ότι τα εργαλεία που, παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στόχο έχουν τη διευκόλυνση τη συλλογή των υπογραφών και τίποτα παραπάνω. Οπότε οι δύο οργανωτέ οι ίδιοι θα πρέπει να το θέσουν σε εμπορία και να δημοσιοποιήσουν τι πρωτοβουλίε. Εμεί προσφέραμε τεχνική αρρωγή για να βελτιστοποιήσουμε την προετοιμασία και τη χρήση της ε, νέας αυτής διαδικασία. Επίση, υπάρχουν ισχυρισμοί ότι το ε, λογισμικό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής δεν είχε δοκιμαστεί επαρκώ. Αυτό δεν αληθεύει. Έγιναν δοκιμέ, ε, ακόμη σε επίπεδο ε, μονάδας, έγιναν δοκιμές ευαισθησίας του συστήματος και φυσικά επιδέχεται βελτιώσει, χρησιμοποιείται πάντα κοινοτική προσέγγιση και έχουν αναλυφθεί βήματα. Επίση, ένα σεμινάριο για λογισμικό ανοιχτή πηγή open source έχει αρχίσει ε, με συμβολές ε, από εξωτερικούς φορείς ε, και προς το παρόν δύο εταιρείε έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για να μετάσχουν στη διαδικασία. Έμεσα είμαστε σε επαφή φυσικά και με τους πολίτες. Η πιο νομοποιημένη αν θέλετε ανησυχία που εκφράστηκε είναι ότι οι, όσοι ανέπτυξαν το λογισμικό δεν υποστήριξαν στη συνέχεια τη διαδικασία. Αυτό δεν συνδέεται όμως με την πλατφόρμα συλλογής υπογραφών της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Το νομικό πλαίσιο δεν επαρκεί. Η νομοθετική πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπει σε όλου του πολίτε να ασκήσουν τα δικαιώματα του όπου και αν διαμένουν. Όμω ο κανονισμό, όπω εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εισήγαγε διάφορε απαιτήσει, διαφορετικέ απαιτήσει μάλλον, για τα δεδομένα ανακράτο μέλο και το Ηνωμένο Βασίλειο ε, και η Ιρλανδία, παραδείγματο χάρη, όταν οι πολίτε του ε, διαμένουν εκτό χώρα δεν μπορούν ε, να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό τη χώρα, αλλά αυτό οφείλεται σε εθνικέ απαιτήσει απαιτήσει. Ε, συμφωνούμε και εμεί ότι αυτό είναι απαράδεκτο ε, και ε, επιμένουμε τα κράτη-μέλη να ελαχιστοποιήσουν στο μέτρο του δυνατού τι απαιτήσει του. Δεν θα έπρεπε δηλαδή να ε, παραγνωρίζουμε τη σημασία αυτών ε, που συνέβησαν ε, κατά το έτος αυτό εφαρμογή γιατί ο στόχος μας είναι να έχουμε μια ευτυχή έκβαση με αυτή τη νέα πρωτοβουλία. Κλείνοντας, θα έλεγα ότι το Κοινοβούλιο έχει ένα σημαντικότατο ρόλο, διότι ανέλαβε εξ αρχή σε δέσμευση, ούτω ώστε να τελεσφορήσουν οι προσπάθειές μας. Αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΔΕ ότι όταν εντοπίζονται δυσλειτουργίες του συστήματος, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κοινού στόχου. Θέλουμε επανασύνδεση με του πολίτε Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή συμμετοχή στο δημοκρατικό βίο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοβουλία των πολιτών είναι πάρα πολύ σημαντική προσθήκη ε, στα πιο παραδοσιακά μέσα και υποδομέ συμμετοχική δημοκρατία και συνιστά εναλλακτική λύση για του πολίτε ε, που θέλουν ε, να εμπλακούν άμεσα στον ευρωπαϊκό βίο και να είναι σε άμεση σύνδεση με τα θεσμικά όργανα τη Ένωση. Σα ευχαριστώ και ελπίζω να διευκρίνησα κάποια επιμέρου σημεία. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Ακολουθούν πολιτικές ομάδες από το ΕΛΚ η κυρία Κάμπριερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το 2013 έχουμε δύο επαιτίους. Δύο χρόνια ε, ε, ζωής για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία και ένα έτος πρακτικής εφαρμογής αυτής. Ποιος είναι σήμερα ο απολογισμός. Η συμμετοχική δημοκρατία κυριαρχεί ε, στη δημόσια συζήτηση 1,5 χρόνο πριν τις ευρωεκλογέ. Αυτό είναι ένα μήνυμα που δίνουμε εμείς στις κοινωνίες μας επιμένοντας ε, στις αρχές μας και προσπαθώντας να έρθουμε πιο κοντά ε, στους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτή η πρωτοβουλία είναι σημαντική και χρήσιμη για τους πολίτες για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε και να έχει αποτελέσματα με διαφάνεια και να στεφθεί με επιτυχία. Η πρωτοβουλία αυτή έχει πολλά θετικά. Είναι μια πρώτη υπερεθνική πλέον πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μπορεί να ε, διορθώνει τα σφάλματα ε, που διαπράττουμε κατά τη διάρκεια των ε, νομοθετικών μας εργασιών. Είναι θετική λοιπόν ε, αυτή η διαδικασία. Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες ε, και σε σύγκριση με τις καταγγελίες προς το διαμεσολαβητή ή τις αναφορές, έχει προστιθέμενη αξία η πρωτοβουλία αυτή και σε αντίθεση με τα δημοψηφίσματα όπου η απάντηση είναι μόνο ναι ή όχι, μέσω της πρωτοβουλίας αυτής μπορούν οι πολίτες να κάνουν προτάσεις για να διορθώνουν τα δικά μας σφάλματα. Θα πρέπει λοιπόν να ε, υλοποιηθεί αυτή η προσπάθεια ε, τη πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Αντιμετωπίζουμε πολλά εμπόδια. Ο κόσμο δεν το γνωρίζει αυτό το μέσο που έχει στη διάθεσή του. Πρέπει να το προβάλλουμε περισσότερο, να το διαφημίσουμε για να ξέρουν οι πολίτε πώ θα προσπίσουν τα συμφέροντά τους. Πώς θα το κάνουμε αυτό, πώς μπορούμε να κάνουμε ευρύτερε εκστρατείε, καμπάνιες ενημερωτικέ, πώς μπορούν να μαθαίνουν οι πολίτες για αυτή την πρωτοβουλία και να την κάνουν κτήμα τους. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν τη διαδικασία. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ε, ανάμεσα ε, στις προσδοκίες ε, των Ευρωπαίων πολιτών και στην νομοθεσία που εκ των ενστέρων εμείς εγκρίνουμε. Θα πρέπει να τροποποιηθεί και η διαδικασία. Η Επιτροπή ε, Αναφορών και διάφορες εισηγητές τη συγγνώμη, έχουν προτείνει τροπολογίες. Δεν είναι πάντα εύκολα όλα αυτά να υλοποιούνται. Χώρα η βελτίωση, η διαδικασία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν βέβαια στο πλευρό μα. όταν χρειάστηκε να ληφθούν ad hoc και προσωρινά μέτρα, αλλά θα πρέπει να παρακολουθούμε τα τεχνικά στοιχεία και ιδιαίτερα αυτό το θέμα του λογισμικού. Επίσης, Υπάρχει μια προθεσμία 12 μηνών για τη συλλογή υπογραφών. Ορισμένε πρωτοβουλίε είναι εκπρόθεσμε. Θα κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχουν όλοι οι ίσε ευκαιρίε στην πρόσβαση. Θα πρέπει να είναι λοιπόν συγκεκριμένε πάντα οι πρωτοβουλίε και τελικά να καταλήγουν σε νομοθεσία. Ο δικό μα ρόλο ποιο είναι σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ χρήσιμοι στους πολίτες, διοργανώνοντας ακροάσεις και άλλες δραστηριότητε, πάντα σε στενή συνεργασία, χέρι με χέρι, για να τους βοηθούμε και να επιμείνουμε στη βαθύτερη ουσία αυτής της πρωτοβουλίας. Ο κύριος Γκερέρος Σαλόμου, σοσιαλιστές, για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει νομίζω ευρεία συνένεση στο να θεωρήσουμε ότι μία από τις μεγάλες καινοτομίε της συνθήκης της Λισαβόνα ήταν το να αναγνωριστεί στους πολίτες η ικανότητά τους να να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες των πολιτών. Σε αυτή τη βάση, η δουλειά της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου για την έγκριση της αντίστοιχη ε, νομοθεσίας νομίζω ήταν ικανοποιητική, σχετικά ταχεία και ούτως ή άλλως πολύ θετική σε σχέση με αυτά τα δικαιώματα των πολιτών. Δεν υπήρξε καμία αντίσταση στο Κοινοβούλιο ως εκπρόσωπο της ε, αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας σε αυτή την πρωτοβουλία. Κάθε άλλο, πάντοτε θεωρήσαμε ότι αυτό πετέλεσε ένα εμπλουτισμό της δυνατότητές μας για αντιπροσώπευση των πολιτών. Θα έπρεπε να κάνουμε μια αναθεώρηση το 2015. Η αλήθεια είναι όμως ότι είμαστε υποχρεωμένοι να την κάνουμε από τώρα, Άμεσα δηλαδή, επειδή ένα έτος μετά από την εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας, καμία από αυτές τις πρωτοβουλίες δεν έχουν υλοποιηθεί. 30 κατατέθηκαν, 14 συνεχίζονται και υπάρχουν προβλήματα που βεβαίως φρενάρουν την εφαρμογή τους. Θα μπορούσαμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για τα θέματα τα οποία ενδιέφεραν τους πολίτες είναι θέματα με ψηλό κοινωνικό περιεχόμενο. Έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής, με το περιβάλλον, έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία, με την έρευνα, με τα δικαιώματα. Γι' αυτό ακριβώς είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν υπήρξε εκ μέρου του λόμπι της αγοράς μια χειραγώγηση αυτών των πρωτοβουλειών. Όμως η Κομισιόν μόλις αναφέρει και συμφωνούμε όλοι από αυτό ότι υπάρχουν τεχνικά και νομικά και υλικά προβλήματα. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να ζητήσει από το Συμβουλίο να μειώσει τα προβλήματα τα οποία βρίσκονται στα χέρια των χωρών μελών. Κυρίως αναφέρθηκαν η να αναγνώριση των υπογραφών πολιτών που ζουν εκτός χώρας και νομίζω ότι Πρόεδρε υπάρχει αρκετός ευροσκεπτικισμός. Θα πρέπει να δώσουμε λοιπόν στους πολίτες τη δυνατότητα να νιώσουν Ευρωπαίοι και μετέχοντες της νομοθετικής διαδικασίας. Ευχαριστώ. Ο κ. Ελουάρτ και τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε υπό τη Λισαβόνα αυτή η πρωτοβουλία θεωρήθηκε ως κάτι το οποίο γεφύρωνε το δημοκρατικό χάσμα, ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο έβαζε τους πολίτες στο κέντρο της Ευρώπης. Νομίζω ότι αν δούμε τη συμμετοχή των πολιτών θα δούμε πού βρίσκονται τα προβλήματα. Για παράδειγμα, είδαμε στην Ιρλανδία ότι το 86% των πολιτών είχαν ακούσει για αυτή την πρωτοβουλία, ενώ το 70% θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν. Η πρωτοβουλία των πολιτών, το ίδιο λοιπόν εργαλείο αυτό που σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει το δημοκρατικό έλλειμμα και για να, για να εμπλέξει τους πολίτες στη δικασία του εκδημοκρατισμού της Ευρώπης βρίσκεται μακριά από το να του συνειδητοποιήσει σε σχέση με την διαδικασία λήψη αποφάσεων στην Ευρώπη. Το γεγονό ότι 70% των πολιτών θα ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν αποδεικνύει ότι υπάρχει βούληση για πραγματική εμπλοκή στη δικασία λήψη αποφάσεων. Όμω πρέπει να πούμε ότι οι πολίτε θέλουν να συμμετέχουν, θέλουν να συμβάλλουν και θέλουν να ακούσουν η φωνή του. Το γεγονό λοιπόν ότι αυτέ οι πρωτοβουλίε λήφθηκαν αποδεικνύει το γεγονό ότι έχει μεγάλο δυναμικό αυτό το εργαλείο σε σχέση με τους ομιχοί των πολιτών. Θα πρέπει εμείς να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες για τη συμμετοχή των πολιτών ώστε να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη των πολιτών μαζί με τους πολίτες. Ε, μια από τις κύριες επικρίσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι δεν επικοινωνεί με τους πολίτες της και η άλλη είναι ότι η νομοθεσία γίνεται από, κάτω προς, από πάνω προς τα κάτω. Αυτή η πρωτοβουλία λοιπόν των ε, πολιτών, αν εφαρμοστεί με το σωστό τρόπο, θα αποτελεί το εργαλείο για την συμμετοχή των πολιτών. Όμως, παρουσιάζει και υπερβολική γραφειοκρατία και δισκαμψία τα διοικητικά κριτήρια νομίζω ότι είναι προβληματικά. Υπάρχουν διάφορα παράπονα για θέματα έλλειψης διαφάνειας και ε, παραδεκτού. Η πρωτοβουλία των πολιτών δεν θα πρέπει να αποτελεί χάσιμο χρόνο. Θα πρέπει η δικασία να επιταχυθεί και θα πρέπει τα προβλήματα με τη συλλογή των υπογραφών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με το ταχύτερο δυνατό και πρακτικό τρόπο, ώστε να αποτελέσει αυτή η πρωτοβουλία ένα εργαλείο σωστό για τους πολίτες υποστηρίζω πλήρως την ιδέα ότι θα πρέπει να πληροφορούνται και ενημερώνται καλύτερα οι πολίτε 27 και τώρα 28 χώρε. Θα πρέπει επίση να δούμε τι γίνεται με τα θέματα εθνικότητα και κατοικία των πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει η απαραίτητη υποστήριξη προ αυτή την ε, πρωτοβουλία που αποτελεί ένα σημείο κλειδί τη ε, Λισαβόνα, ώστε να διασφαλίσουμε την πλήρη συμμετοχή των πολιτών και να μην μείνει στο γράφει τελικά αυτή η πρωτοβουλία. Τέλος, Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άμεσα προς την Κομισιόν. Γιατί δεν έχουμε μια πρωτοβουλία ηθαγένειας ή πολιτών για την ε, ενιαία έδρα των ευρωπαϊκών εργών. Νομίζω κάτι τέτοιο είχε προταθεί και θα ήθελα να ακούσω σας. Ευχαριστώ. Κύριε μια γαλάζια κάρτα του κυρίου Τηλεφωνεί στο μεταξύ. Ναι, το κύριο Μακμίλαν. Ναι, πολύ σύντομα. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Έλγορ, δεν θα συμφωνούσε ότι είναι λυπηρό στις ε, διαπραγματεύσεις για την πρωτοβουλία των πολιτών. Ένα κράτος μέλος επέμενε να αποκλειστεί οποιαδήποτε πρωτοβουλία ε, που θα αφορούσε ε, την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κυρία Μάλστρομ όταν ε, ήταν ε, ευρωβουλευτής, έκανε μια αναφορά για την ενιαία έδρα στις Βρυξέλλες που έλαβε 1,27 εκατομμύρια υπογραφές. Και τώρα η κυρία Ματσόνη και ο κύριος Σούλτς τα μπλοκάνουν Μάλιστα, ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό και θα ήθελα να το απαντήσει η Επίτροπος στη δευτερολογία της. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Κιέφνερ έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. liebe Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι μια μεγάλη χειρονομία, μια προσφορά μας προς τους πολίτες Ευρώπης. Τους είπαμε, η Ευρώπη αυτή δεν είναι η Ευρώπη των θεσμικών οργάνων ούτε των κυβερνήσεων είναι και η Ευρώπη και κυρίως και πρώτα απ' όλα η Ευρώπη των πολιτών, η δική μας Ευρώπη, η δική σας Ευρώπη. Ανακατευθείτε, κάντε προτάσεις, συμμετέχετε, πείτε μας τα μελήματά σας, τις ανησυχίες σας. Αυτή ήταν μεγάλη προσφορά ε, με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και ε, είμαι ακόμη υπερήφανο που επέτυχε αυτή η προσπάθεια και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν. Να θυμίσω ότι αυτό ανάγεται σε μια πρωτοβουλία των ίδιων των πολιτών. Περισσότερη δημοκρατία λεγόταν από τη Γερμανία, η ΜΚΟ, η Eurotopia, ε, το Ινστιτούτο για την Ευρώπη, Δημοκρατία για την Ευρώπη, διάφορες οργανώσεις και ε, πάρα πολύ ε, ενεργά και στρατευμένα μέλη της συντακτική συνέλευσης, αν θυμάστε, το είχαν αναλάβει αυτό. Και στη συνέχεια ε, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζήτησαν, θα τα θυμάστε αυτά, ήταν μεγάλες οι συζητήσεις και μακρές και σήμερα τι λέμε, ότι αυτή η μεγάλη υπόσχεση προς τους πολίτες έχει εκπληρωθεί μόνο εν μέρη. Σε εμά εναπόκειται αν θα καταφέρουμε πλήρως να την τηρήσουμε ή να την αφήσουμε ημιτελή. Είναι σαφές όταν δημιουργείς για πρώτη φορά ένα νέο μέσον, ε, είναι αχαρτογράφητα ύδατα. Είναι ε, σαν ένα ε, παιδί που μπουσουλάει και σιγά σιγά σηκώνεται και αρχίζει να περπατάει. Ε, δεν μπορεί και να τρέξει αμέσως γιατί είναι πάρα πολύ βαριά τα πόδια του και θα πρέπει όλα αυτά τα βαρύδια να φύγουν το ένα μετά το άλλο. Βαρύδι πρώτο. Οι περισσότεροι πολίτες στην Ευρώπη δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει αυτό το μέσο και το εργαλείο στα χέρια τους. Πριν τη θέση σε ισχύ, Είχα απευθυνθεί στον πρόεδρο Σουλ, στον πρόεδρο Μπαρόσο και στον πρόεδρο Φαρόμπαϊ και τους πρότεινα να βγουν από κοινού ενώπιον των πολιτών και να το ε, εξαγγείλουν. Αρχίζει μια νέα εποχή. Θέλουμε να ακούμε και τις δικές σας προτάσεις. Δεν θέλουμε μια Ευρώπη που να αποφασίζει και να ακούγεται από πάνω προς τα κάτω. Θέλουμε να είμαστε και μια Ευρώπη που να ακούει και να εισακούει τους πολίτες. Αξιοποιήστε το. Δεν έχει χαθεί ακόμα η ευκαιρία αυτή. Είμαστε στο έτος των Ευρωπαίων πολιτών και θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και λογικό να αξιοποιήσει τη δυνατότητα αυτή η Κομισιόν αλλά και τα τρία θεσμικά όργανα να βγουν από κοινού και να το εξηγήσουν στους πολίτες και να το διαφημίζουν στους πολίτες. Ακριβώς αυτή τη χρονιά που είναι το έτος του Ευρωπαίου πολίτη να τους εξηγήσουμε ότι οι πολίτες σας χρειαζόμαστε, συμμετέχετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δίνει τόσα λεφτά για τη διαφήμιση, ακόμα και για τις ευρωεκλογέ, παρόλο που το έχουν καταλάβει οι πολίτες, εν πάση περιπτώσει, ότι έχουμε εκλογέ. Ε, το ακούνε από τις τηλεοράσεις, από τα μέσα ενημέρωσης, ε, από τις αφήσει δεν χρειάζεται να κάνουμε εμεί διαφήμιση γι' αυτό. γιατί την πρωτοβουλία των πολιτών πρέπει όμω. Και μετά υπάρχουν και πολλέ τεχνικέ δυσκολίε. Ουδέποτε το λογισμικό είχε δοκιμαστεί στο παρελθόν. Χάσαμε μήνε γιατί δεν μπορούσαν να συλλέξουν ηλεκτρονικά υπογραφέ. Τώρα έχει βρεθεί μια λύση ad hoc για περιορισμένη ε, και σε αριθμό και σε χρονική διάρκεια ε, εφαρμογή. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα όπου όλες οι πρωτοβουλίες να μπορούν να υποβάλλονται, να παρακολουθούν οι πολίτες και μια πλατφόρμα που να είναι τελείως δωρεάν για τους πολίτες και απλή στη χρήση. Και κατά τα άλλα πολλά προβλήματα Ε, δεν έχουν να κάνουν με το λογισμικό αλλά με την περιπλοκότητα του ίδιου του κανονισμού και όλες αυτές τις απαιτήσει που βάζουν τα κράτη-μέλη για την επιστοποίηση. Μα δεν μπορούμε επιτέλους να ε, το εναρμονίσουμε αυτό. Όνομα, διεύθυνση, υπογραφή. Τελείωσε σε όλα τα κράτη-μέλη και σε λιγότερο από τρία χρόνια μπορούμε ανα πάσα στιγμή να το μεταρρυθμίσουμε και το Κοινοβούλιο είναι ε, γι' αυτό πάντα πρόθυμο. Ευχαριστώ κύριος Βλάσακ, νομίζω ότι απουσιάζει. Οπότε, ο κύριος Μπάτεν, για 1,5 λεπτό. Ε, thank you very much, Madam President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μια άσκηση δημοσίων σχέσεων ε, για να καλύψουμε την μη δημοκρατική Ευρώπη προτάσσοντας αυτό το δημοκρατικό εργαλείο. Ο Άμπραχαμ Λίνκον είπε ότι είναι η κυβέρνηση των ανθρώπων από τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν όμως τέτοιοι εκείνοι άνθρωποι στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει πολιτική ταυτότητα με την οποία να μπορούν να ταυτιστούν. Άρα γνήσιο δημοκρατικό σύστημα είναι ανέφικτο ούτως ή άλλως να συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται για μια δημοκρατία των κρατών εθνών όπου οι πολίτες ε, θα πρέπει να αναγνωρίσουν μια κοινή πολιτική ταυτότητα. Αυτό χρειάζεται. Όμως η δημοκρατία έχει διαφορετικές εκφάνσεις και υποδομές ε, ανάλογα με τη χώρα. Όμως ε, για να είναι γνήσια η δημοκρατία χρειάζεται ένα ενιαίο χαρακτηριστικό. Όχι μόνο να, μπορεί να εκλέξει ο λαός την Ευρώπη αλλά και να αποπέμψει την κυβέρνηση. Να ένα πράγμα που δεν μπορούμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένωση. Δεν επιλέγουν οι άνθρωποι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι η κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί να απολύσει ως εκ τούτου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε όταν κάποιοι ισχυρίζονται ότι λειτουργεί αισίως η δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς θεωρούμε ότι καταστρέφεται. Στο δυτικό κόσμο και κυρίως στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε αποσύνδεση των κυβερνήσεων από τους πολίτες, επιβάλλονται ανεπιθύμητες πολιτικές, όπως παραδείγματος χάρη μαζική και μη ελεγχόμενη μετανάστευση απαγόρευση ανόητες ε, ε, περιβαλλοντικές ε, πολιτικές που καταστρέφουν και την οικονομία των κρατών. Η πρωτοβουλία του να αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν το μόνο λογικό και το UKIP αυτό είχε αποφασίσει και προτείνει αυτή τη γραμμή. Ευχαριστούμε ο Σόλτ, ένα 1,5 λεπτό. Στο... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, υπέγραψα την προφορική ερώτηση διότι θεωρώ ότι είναι σωστέ οι ερωτήσεις που σας έχουν υποβληθεί, άλλωστε το δείχνει και η σημερινή συζήτηση. Ε, θα πρέπει σύντομα να αρθούν τα εμπόδια και δυναμίες που έχουν διαπιστωθεί. Φαίνεται ήδη από σήμερα ποιο είναι το βασικό θέμα που πρέπει να διορθωθεί. Τα μεγάλα γραφειοκρατικά εμπόδια πρέπει να μειωθούν και το ίδιο το μέσο να γίνει πολύ πιο ευέλικτο. Ονομάζεται πρωτοβουλία των πολιτών Και δεν ήταν ο στόχο να υπάρχει μεγάλη οργάνωση ΜΚΟ για μπορούν να φτάσουν μέχρι την Κομισιόν ή μέχρι το Κοινοβούλιο. Δεν λειτουργούν έτσι οι κοινωνίε μα. Συμμετοχή, ε, ανάμειξη στα κοινά θα πρέπει να μπορεί κάθε πολίτη να έχει τη δυνατότητα. Και εμεί θα πρέπει να βοηθήσουμε. Γιατί να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Γιατί να μην συνδέσουμε την πρωτοβουλία των πολιτών με τη δική μας κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Έχουμε και τις ακροάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θα πρέπει ε, να χάνονται οι πρωτοβουλίε που δεν θα έχουν συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών, να χρησιμοποιούνται και να ε, ως ε, αναφορές. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Αυτό τον καιρό τρέχει η πρωτοβουλία Right to Water, δικαίωμα στο νερό, για την ε, καταπολέμηση της ιδιωτικοποίησης των υδάτων. Πάνω από ένα εκατομμύριο έχει συλλέξει και σε πέντε κράτη-μέλη την απαρτία επίσης. Στην Ιταλία δεν έχει συμβεί αυτό, αλλά πριν από δύο χρόνια μάζεψαν ε, υπογραφές πάνω από 1,4 εκατομμύρια. Αυτό θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε και να πούμε ότι από κοινού αναλαμβάνουμε κάποια δράση. Να διοργανώσουμε μια νέα πρωτοβουλία πολιτών. Ευχαριστώ κύριος ε, Μέλτσερ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι πλέον γνωστή, έχει τεθεί σε ισχύ πριν από ένα χρόνο. Θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους πολίτες να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και στην νομοθεσία ταυτόχρονα με διαφάνεια, με εγκύτητα στον πολίτη. Αλλά μέχρι τώρα τι μας δείχνει η εμπειρία. Δυστυχώς δεν κατάφερε αυτό να γίνει ουσιαστική πραγματικότητα. Ε, πολλοί πολίτες ε, καταγγέλουν για τη γραφειοκρατία, τα τεχνικά προβλήματα και το υψηλό ή απαγορευτικό κόστος. Οι ε, Global 2000 της Αυστρίας μου γράφουν ότι ένα χρόνο μετά Ε, την ανάληψη πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση της πυρηνικής ενέργειας ε, πρέπει να αποσύρει την πρωτοβουλία λόγω ε, τεχνικών, γραφειοκρατικών προβλημάτων και μεγάλων εμποδίων ως προς τη δαπάνη. Αυτά λέγουν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι εύκολη η πρόσβαση, φιλική προ το χρήστη για να ανταποκρίνεται στον αρχικό στόχο ε, της πρωτοβουλία των πολιτών. Αυτό που θέλουμε δεν είναι πρωτοβουλία, είναι η συμμετοχή των πολιτών. Ε, στην αρχή είπα ότι είναι επικίνδυνο να δίνουμε στους πολίτες δυνατότητα ε, συναπόφασης ή μάλιστα να του την προβάλλουμε και ως κίνητρο και ως πρόφαση που τελικά δεν τη διαθέτει. Ε, αυτό ε, δεν δίνει μεγαλύτερη αξιοπιστία στην πρωτοβουλία. Θα πρέπει να σκεφτούμε ε, μήπως οι ε, ε πρωτοβουλίες που ευδοκιμούν θα πρέπει να οδηγούν σε αυτόματη δράση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τέσσερα λεπτά ο κύριος Μπέκερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Ένα έτος Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών είναι αφορμή για συγχαρητήρια, κυρίως τους τόσο άριθμους πολίτες που σε όλη την Ευρώπη ε, έχουν συμμετάσχει στο πρώτο υπερεθνικό εργαλείο άμεσης δημοκρατίας. 14 πρωτοβουλίες έχουν κατατεθεί ήδη. Και χαίρομαι που ως Αυστριακός ε, οι τέσσερις προέρχονται από την Αυστρία υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, παρακολούθησαν αυτό το εργαλείο όχι μόνο από την αρχή αλλά το υποστήριξαν ουσιαστικά ε, για την ε, επιγραμμική συλλογή υπογραφών. Συγγνώμη. Η πρωτοβουλία πολιτών σημαίνει όμως και μία κριτική ενδιάμεση αξιολόγηση, έναν απολογισμό για να δούμε πού μπορούν να γίνουν αλλαγές και βελτιώσεις. Το βασικό πρόβλημα αυτού του νεοπαγούς μέσω στην Ευρώπη είναι βεβαίως η ε, γνώση των πολιτών. Και ξέρετε δεν είναι αυτό μόνο ευθύνη και καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι μεν αλλά και των κρατών μελών. Μέχρι τώρα δεν έχουν δραστηριοποιηθεί. Ε, μου λείπει αυτή η συμμετοχή τους. Και άλλα δεινά είναι αυτή η ηλεκτρονική συλλογή ε, ε, υπογραφών. Υπάρχουν τεχνικά και γραφειοκρατικά εμπόδια. Μία ιδέα που αξίζει να ακολουθηθεί είναι να υπάρχει ένα λογισμικό έτοιμο προς χρήση και να διατίθεται σε όλους τους ενδιαφερομένους. Εχθές πήρα πέντε email, κυρία Επίτροπε, και θα τις έχετε λάβει κι εσείς, ομάδες πολιτών ζήτησαν 12 μήνες για τη συλλογή των υπογραφών από τη στιγμή που θα ε, ανέβει στο διαδίκτυο η πρωτοβουλία. Νομίζω είναι πολύ πρακτική αυτή η πρόταση γιατί είναι πραγματική 12 μήνες ε, για τη συλλογή των υπογραφών. Δηλαδή η αντίστροφη μέτρηση να αρχίζει από τη στιγμή που θα εγκριθεί και θα πιστοποιηθεί η πρωτοβουλία. Να αναφέρω όμως και ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ προσωπικά και με αφορά. Αυτό το πρώτο έτος Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας ε, Πολιτών θα πρέπει και είναι θεμητό να αναρωτηθούμε για ορισμένε δραστηριότητες. Τι εννοώ, υπάρχει μια πρωτοβουλία ε, που ε, ξεπέρασε ως πρώτη το ένα εκατομμύριο για το νερό. Είναι αυτή η ιστορία με τα ύδατα και δεν τυχαίο που ε, έχει κινητοποιηθεί από μια ε, ομάδα λαϊκιστών. Έγινε λόγος για ε, αναγκαστική ιδιωτικοποίηση του νερού που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό απεδείχθη ασφαλμένο. Σε αυτή τη διαδικασία όμως της εκστρατεία και της καμπάνιας είμαστε υποχρεωμένοι να διαπιστώσουμε ότι οι βασικοί υποκινητές αυτής της πρωτοβουλίας και αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό τα ευρωπαϊκά συνδικάτα σίγουρα δεν ήταν ο αποδέκτης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα είναι συγκροτημένος φορέας συντεταγμένης πολιτείας, δεν είναι ε, πρωτοβουλία πολιτών, δεν είναι ομάδα πολιτών το συνδικάτο. Γι' αυτό ε, νομίζω ε, θα ήταν σωστό το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα να το ξανασκεφτεί και στο μέλλον να αποσύρει αυτή τη δράση του και να μην συμμετέχουν σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Είναι ένα εργαλείο αυτό άμεσης δημοκρατίας, όχι της συντεταγμένης πολιτείας. Το διαστρεβλώνουν, το σφετερίζονται και το χρησιμοποιούν για λάθος τρόπο. Δεν θέλω εγώ να ζω σε μια Ευρώπη χωρίς συνδικάτα αλίμονο, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ε, να μην ε, σφετεριζόμαστε. Αυτό είναι δικαιώματα πολιτών, όχι τα δικαιώματα των συγκροτημένων, ε, συντεταγμένων οργάνων της πολιτείας. Είμαστε όλοι περήφανοι για την πρωτοβουλία αυτή, αλλά θα πρέπει να βελτιωθεί και να αξιοποιηθεί στο έπακρο. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκουρμά για δύο λεπτά. Thank you very much, dear Vice President. Ευχαριστώ πολύ. Αντιπρόεδρε, ήμουν συνεισηγήτρια για αυτό το πολύ σημαντικό εργαλείο και χαίρομαι πάρα πολύ που το συζητάμε τώρα. Η ΠΕΠ αποτελεί ένα παραστατικό εργαλείο για τη δημοκρατία και επιτρέπει στους πολίτες να ακουστούν την εποχή και τον καιρό που χρειάζεται περισσότερο. Ο αριθμός των πρωτοβουλειών που έχουν καταβληθεί μέχρι τώρα και το γεγονό ότι παρουσιάζουν τόμε ιδέε με κάνει ένα Νομίζω ότι πραγματικά οι Ευρωπαίοι πολίτε άρχισαν να διακρίνουν την προσθέμενη αξία του εργαλείου. Παρ' όλα αυτά, η θετική αυτή εξέλιξη δεν θα πρέπει να αποκρύπτει τι τεχνικέ δυσκολίε που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτέ μέχρι τώρα και τι προκλήσει που απομένουν. Βεβαίω, είναι αλήθεια ότι με το νομοθετικό έργο για αυτό το εργαλείο είχαμε μπει σε χαρτογράφητη, αγιογράφητη περιοχή και έχουμε προβλήματα ιδιαίτερα όσον αφορά τους servers για την online συλλογή των υπογραφών. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια βιώσιμη λύση και το ίδιο ισχύει και την ανέβρεση ισορροπίας μεταξύ προστασίας των δεδομένων και της φιλικότητας προς το χρήστη. Ξέρω ότι κάποιοι ζητούν αναθεώρηση του κανονισμού, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς Χρειαζόμαστε μια πλήρη αξιολόγηση πριν να ξεκινήσουμε μια τέτοια διαδικασία. Καλωσορίζω τις προσπάθειες που έκανε η Κομισιόν μέχρι τώρα, όπως η απόφαση η απόφαση του να επεκταθούν στη 12η περίοδο μετά από τι πρώτε πρωτοβουλίε, ώστε να αντιμετωπιστούν τα τεχνικά προβλήματα. Και θέλω να υπογραμμίσω και την σημασία τη ίση μεταχείριση. Θα πρέπει να γίνουν πολλά βεβαίω για την αναθεώρηση μέχρι το 2015 από του διοργανωτέ και από την κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει βεβαίω να ληφθεί υπόψη οι εμπειρίε που υπάρχουν, ώστε να γίνει η συλλογή των υπογραφών online πιο ανοιχτή και να υπάρχει μια αποκεντρωμένη διαδικασία. Επίσης θα πρέπει να ξαναχρησιμοποιήσουμε, να μειώσουμε όσο γίνεται το κόστος ε, της ε, ΠΕΠ γιατί πάρα πολλοί πολίτε δεν έχουν ακόμα γνώση της ύπαρξη του εργαλείου αυτού και αυτό είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των ε, γραφείων πληροφοριών. Θυμάμαι ότι υπήρξε περίπτωση μιας ε, χώρας μέλους που μπλόκαρε τη συλλογή των, ε, ε, των υπογραφών για κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει πλήρης ίση μεταχείριση για δημοκρατική διαφάνεια. Εδώ ευχαριστώ. Ναι, απευθύνομαι στους πολίτες που παρίστανται σήμερα ως ακροατές. Θα ήθελα να σας πω ότι η ευκαιρία είναι πολύ καλή αυτή, πολύ σημαντική και θα πρέπει να την λάβουν υπόψη σοβαρά και να ακούσουν προσεκτικά τις αναλύσεις που γίνονται. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Ρινάλντι για δύο, δύο μισή λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητή Σεσίλια, αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για τα λίγα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για μια άμεση σχέση μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Όχι μόνο στα πλαίσια του έτους των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά σε μια περίοδο όπου η αξιοπιστία της ΕΕ στην κοινωνία μας βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά. Δεν μας το λέει αυτό η Eurostat, αλλά η καθημερινή εμπειρία που έχει ο καθένας από εμά στις επαφές τους με τους πολίτες. Τώρα η πρωτοβουλία αυτή, η ΠΕΠ, αποτελεί ένα όπλο που αν χρησιμοποιηθεί σωστά θα μπορούσε να είναι θαυμάσιο. Εγώ ήμουν από τους προωθητές μας με άλλους μιας πρώτης ε, πρωτοβουλίας που ζητούσε ένα πλουραλισμό στην ενημέρωση. Το Κοινοβούλιο την υιοθέτησε, φτάσαμε σε μια ιστορική ψηφοφορία 334 ε, ψήφι υπέρ, 334 κατά ε, ισοπαλία, ισοψηφία που έκανε την πρωτοβουλία αυτή να καταπέσει. Αλλά τι ωραία θα ήταν να δίνουμε ειδήσει και νέα στους Ευρωπαίους πολιτές μέσω της ΠΕΠ και της συλλογής των υπογραφών που χρειάζεται ένα πρόβλημα όμως που δεν, που, δεν μπορέ... που δεν μπορέσαμε να λύσουμε στα εσωτερικά των θεσμικών οργάνων θα μπορούσε να βρει μια λύση μέσω αυτής της πρωτοβουλίας για θέματα που αφορούν τον πλουραλισμό και που είναι στον ίδιο το πυρήνα των αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κάνουμε λοιπόν για να βοηθήσουμε εμείς αυτή την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Θέλω να πω ότι η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ καλή επειδή ε, φτάνει ακριβώς ένα έτος μετά από την θέσπισή της. Και είναι αναγκαίο να υπάρξει μεταρρύθμιση και αναθεώρηση και υπόθηκε επανειλημμένος. Θα πρέπει να έχουμε ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα όπως αυτό που θα πρέπει να τεθεί στη διάθεση των πολιτών και είναι αλήθεια ότι η χρήση του ενδεχομένως κάποιες φορές να μην είναι πολύ εύκολη για τους πολίτες οπότε εκεί θα πρέπει να παρενεύουμε και από ίδια εμπειρία θα πρέπει να πω ότι υπάρχει σπατάλη χρόνου και χρημάτων που θα πρέπει να αποφευχθεί. Υπάρχουν βεβαίω τεχνικέ προδιαγραφέ για τη συλλογή online που είναι αρκετά περίπλοκε και υπάρχουν και θέματα τα οποία σχετίζονται με τεχνικές και νομικές ε, ε, πτυχέ, όπω η πιστοποίηση των υπογραφών κλπ. και άλλα θέματα τα οποία ήδη έχουμε κοινοποιήσει στην Κομισιόν. Αλλά θα πρέπει να δούμε κυρίω τι έχουμε κάνει όλοι μα, εμεί οι βουλευτέ, για να προωθήσουμε αυτό που αποτελεί μια καλή είδηση για του πολίτε. Δηλαδή, κοιτάξτε, υπάρχει αυτό το εργαλείο στη διάθεσή σα. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε η γραφειοκρατία, τα τεχνικά ζητήματα, οι δικοί μα οι ίδιοι περιορισμοί όσον αφορά τι διαφημιστικέ ε, εκστρατείε, να μην ε, υποβαθμίζουν ένα πολύ καλό εργαλείο που προέρχεται από τη Λισαβόνα και ένα θαυμάσιο πολιτικό όπλο. Ευχαριστώ. Ρούκεν, για να Ευχαριστώ. Οι δραστήριοι πολίτες ε, είναι μια, ένας πολύτιμος πόρος. Ε, εργάζομαι στην Επιτροπή Αναφορών και το διαπιστώνω αυτό καθημερινά. Θα πρέπει να έχουμε μια άμεση επιρροή και θα ήθελα ε, να μην γίνει αυτό το εργαλείο πηγή απογοήτευσης. Ε, θέλουμε να συμβάλλουμε στη συζήτηση των ιδεών των πολιτών με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, κυρίως μέσω μιας ομοιόμορφης μεταχείρισης εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει η Επιτροπή Αναφορών να έχει πιο γενικό έργο να είναι δυνατή διοργάνωση ακροάσεων παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, η αρμόδια Επιτροπή θα πρέπει να εκπροσωπείται επίσης αυτές τις ακροάσεις για να έχουμε πραγματικά την αίσθηση ότι επικρατεί σοβαρότητα και μόνο έτσι θα κατοχυρωθεί η συμμετοχή των ε, πολίτων. Ε, ε, θα είναι καταστροφικά τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι τους απατούμε οι πολίτες. Σας ευχαριστούμε, η κυρία Δημαρτίνη, για δύο λεπτά. I'm new here. Πρόεδρε, είμαι νέα βουλευτής και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω διπλά για την ευκαιρία που μου δίνετε να ασκήσω το δικαίωμα για το χρόνο αγόρευσης. Θα μιλήσω Ιταλικά. Η ΠΕΠ είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή τη ε, στιγμή δυσπιστία προς την Ευρώπη. Φαίνεται να αντιμετωπίζει λοιπόν κάποια προβλήματα γραφειοκρατικά και επικοινωνίας, όπως είπε η Επίτροπος και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Να σας δώσω ένα πρακτικό παράδειγμα, μεταξύ άλλων, που αφορά την ίδια μου τη χώρα, την Ιταλία. Η ΠΕΠ για, το, για τα δημόσια ύδατα, όπως υπόθηκε, συνέλεξε σε 9 μήνες πάνω από 20.000 ε, υπογραφέ από τι 34 που χρειαζόταν για την Ιταλία. Ενώ για το ίδιο θέμα σε επίπεδο εθνικού ρεφερέντουμ συλλέχτηκαν το 2011, δηλαδή πρόσφατα, σε λίγου μήνε πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφέ. Αυτή λοιπόν η διαφορά όσον αφορά την επιτυχία μεταξύ τη πρωτοβουλία Μία μόνο χώρα και τη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία δεν εξηγείται παρά μόνο λόγω της ε, δυσκολία στην επικοινωνία και της γραφειοκρατίας. Ξέρω ότι κατατέθηκε μια πρωτοβουλία για την απλούστευση του, της πρωτοβουλίας. Φαίνεται σαν λογοπαίγνιο, αλλά είναι πραγματικότητα αυτό. Μου φαίνεται ότι εδώ έχουμε το παράδειγμα ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι ένα, μια καμήλα που μοιάζει με ένα άλογο, κάτι το οποίο σχεδιάζει ένα ε, γραφειοκράτη. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντεμαρτίνη. Ο του κ. Σισμάνσκι. Ε, Ευχαριστώ. Μαζί με άλλους συναδέλφους από 8 κράτη-μέλη, ε, το κόμμα μου, η ε, Αλληλέγγυα Πολωνία και η ομάδα η αυτή άρχισαν να συλλέγουν υπογραφές για την κλιματική αλλαγή, για να σταματήσει το πακέτο πρωτοβολίας για το κλίμα. Ε, μεγάλη υποστήριξη γνώρισε και την υποστήριξη των συνδικάτων. Το, η ιδέα στη συνθήκη της Λισαβόνα για την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών ήταν σωστή μεν, πλην όμως υπάρχουν δυσκολίες και προβλήματα στην εκτέλεση. Ειδικά σε ό,τι αφορά την ε, επιγραμμική συλλογή υπογραφών και την πιστοποίηση ε, το να γίνεται δεκτή δηλαδή μια τέτοια πρωτοβουλία και δεν κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, διευκολύνει την κατάσταση. Παρά την προσωπική δέσμευση και εργασία ε, μεμονωμένων υπαλλήλων, ε, είναι πολύ βαριά και δύσκολη η διαδικασία. Πώς θα συμμετέχουν οι πολίτες, περιπλοκή τεχνολογία. Είναι μεγάλο και το κόστος, εκτός από τις διοικητικές διαδικασίες. Για να συμπληρώσει κανείς ένα έντυπο χρειάζεται ώρες ολόκληρες. Και δεν υπάρχουν και ε, λεπτομέρειες για το πώς πιστοποιούνται οι υπογραφές που συλλέγονται. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να βρούμε κάποια λύση η οποία να διευκολύνει και να πλουστεύει τη διαδικασία οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δημοκρατική δυνατότητα να ε, προτείνουν τα επιχειρήματά τους και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να τα προωθούν. Είναι κάτι που μας βρίσκει σύμφωνος. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Βίλη Μάγερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα οι μεγάλες συζητήσεις που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση που περιλαμβάνουν πολλές και μεγάλες κινητοποιήσεις και απεργίες και τα λοιπά είναι κατά πόσο θα μπορούσαμε να έχουμε νέο νόμισμα, κεντρική τράπεζα, αν η πολιτική της ε, Ένωσης θα πρέπει να είναι λιτότητας και τα λοιπά. Αυτά είναι τα θέματα που συζητούνται οι πολίτες. Με χαρά θα έπρεπε να έχουν, θα είχαν στη διάθεσή του, θα ήθελαν να είχαν στη διάθεσή του ένα εργαλείο που του επιτρέπει να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Το πρόβλημα λοιπόν που έχουμε είναι ότι το εργαλείο αυτό μπλοκάρει αυτή τη δυνατότητα. Γιατί μπλοκάρει τα θέματα στην ουσία του. Κοιτάξτε, εμεί ω ΓΟΕ είχαμε παρουσιάσει μια πρωτοβουλία σε σχέση με την δημιουργία μια δημόσια τράπεζα. Δεν γίνεται αυτό. Μα το αρνήθηκαν. Τον 21ο αιώνα συζητάμε για το κατά πόσο οι πολίτε θα προσεγγίσουν την διαδικασία λήψη αποφάσεω ή όχι. Όλα τα υπόλοιπα είναι παραμύθι. Παραμύθι. Έρχεται λοιπόν ο 21ος αιώνας και οι πολίτες βλέπουν να λαμβάνονται αποφάσεις, να ανακαλώνται αποφάσεις, ε, να γίνονται δεσμευτικά δημοψηφίσματα, αλλά θα πρέπει για αυτούς ακριβώς τους λόγους να ενισχύσουμε τη δυνατότητα των πολιτών να λάβουν μέρος στις συζήτηση και στην ε, λήψη απόφαση. Λήψη απόφαση. Έχει πολύ δρόμο να διανύσει αυτό το εργαλείο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Ο κύριος Μπουλάν, τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ. Η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών είναι πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των πολιτών, όμως παραλύεται από ε, τις βασικές ατέλειες κάθε γραφειοκρατίας, τα ε, γνωστά γραφειοκρατικά εμπόδια. Ε, το ίμιση ε, ε κρίθησαν απαράδεκτες και σε ένα κράτος μέλος δεν φτάσαμε καν το ένα εκατομμύριο υπογραφές. μετά από πολλές δυσλειτουργίες και ένα χρόνο λειτουργίες θα πρότεινα άρδινα αναθεωρησή του εγχειρήματος, όπως και άλλοι συνάδελφοι, ε, είναι αντιπαραγωγικό αυτό το σύστημα, ισχυρίζονται κάποιοι. Παραδείγματο χάρη ε, στη ΣΥΠΑ κάνουν πρωτοβουλίε πολιτών ε, για το Star Wars. Ε, είναι παράλογο. Επίση, χρησιμοποιείται από συνδικαλιστικέ οργανώσει ή από πολιτικά κόμματα αυτό το εργαλείο ή από κάποιου συναδέλφου. Όπω σα είπα προηγουμένω για την μοναδική έδρα, αυτό αντιβαίνει στι συνθήκε. Μία είναι η έδρα και είναι στο Στρασβούργο. Η πρωτοβουλία πρέπει να παραμείνει στα χέρια των πολιτών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να αντιμάχεται κανεί ε, το νόμο. Όχι, πρέπει να χρησιμοποιείται για να εκδίδεται νομική γνωμοδότηση για κάποιο θέμα. Επίσης ε, πρέπει να είναι στην υπηρεσία όλων ε, και όχι για να αρέσκονται μερικοί. Ε, οι διοργανωτές των πρωτοβουλειών καταδεικνύουν ότι είναι πολυάριθματα εμπόδια αλλά όχι ανυπέρβλητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει υποστήριξη ως προς το λογισμικό αλλά ας απλουστεύσουμε την γραφειοκρατία να έχουμε ένα νέο κέντρο για την συλλογή των υπογραφών και για την πιστοποίηση απλουστεύοντας το θέμα της ταυτοποίησης διότι θέλουμε να αποφύγουμε της απάτης. Όταν εντοπίζεται απάτη, ε, δεν θα πρέπει να θέτουμε να αμφιβόλο την αξιοπιστία της ε, ε, πρωτοβουλίας, αν και είναι επαχθέστερο στη συνέχεια το γραφειοκρατικό έργο. Θα πρέπει να βασιζόμαστε στην επιστοποίηση για να μετρήσουμε την περίοδο και όχι την το, τη στιγμή της συλλογής των υπογραφών. Δεν χρησιμοποιεί σωστά αυτό το σύστημα και οι ετούντες το καταγγέλουν διότι δεν μπορούν ε, να καταθέσουν τις υπογραφές τους. Αν δεν είναι ομοιόμορφοι κανόνε, δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Ταχύτατα πρέπει να δράσουμε για να έχουν εμπιστοσύνη οι κοινωνικοί φορείς μετά από διαβούλευση μαζί τους. Ε, θα ήθελα να τελειώσω με το εξή παράδοξο. Θα πρέπει να έχουμε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για να βελτιωθεί η λειτουργία του θεσμού. Εν μέρη αυτός είναι ε, ο στόχος του ICO 11 που τώρα τρέχει. Θα πρέπει να εντοπίσουμε αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια ε, κατά τη διάρκεια του έτους των Ευρωπαίων πολιτών και ο στόχος ε, θα πρέπει να είναι να μειωθεί ο αριθμός ε, των γραφειοκρατικών κολλημάτων. Ελπίζω να μην αμαυρωθεί η εικόνα αυτού του πολύτιμου εργαλείου συμμετοχής δημοκρασίας και ευρωπαϊκής ηθαγένεια. Σας ευχαριστούμε ο κύριος Μποστινάρου. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Επίτροπε. Είναι η πρώτη επέτειος ε, της λειτουργίας ε, του θεσμού ε, της πρωτοβουλίας των πολιτών ε, όργανο συμμετοχικής δημοκρατίας. Είναι μια αρχή ε, και ήταν μάλλον επιτυχημένη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας μίλησε για το δικαίωμα για νερό για όλους. Συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές και ακόμη δεν έχει κλείσει η διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για τη σύνταξη του κειμένου. Τα δύο τρίτα του κειμένου συγκεκριμένα προέρχονται από το έργο των βουλευτών. Αυτό καταδεικνύει και τη δέσμευσή μας να αυξήσουμε τη συμμετοχή των πολιτών ναι, για να μπορούν να επηρεάσουν και ενδεχομένω και να τροποποιήσουν την κείμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Ο υποφαινόμενος και οι υπόλοιποι συνάδελφοι από την Επιτροπή Αναφορών διαδραματίσαμε πολύ σημαντικό ρόλο για την προώθηση αυτού του εργαλείου συμμετοχικής δημοκρατίας. Θα ήθελα να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσέξει τους κινδύνους ε, που ελοχεύουν, δηλαδή να χρησιμοποιηθεί αυτό το εργαλείο σε κάποια κράτη-μέλη για λόγους ε, έθνη ε, κόφρονης προπαγάνδας, για να επιτρέψουν στους πολίτες να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Ευχαριστούμε κύριε Άντερσον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι η πρωτοβουλία αυτή είχε λιγότερο αντίκτυπο από αυτό που θα ήθελαμε. Εγώ συμμετείχα σε πολλές δικασίες και εκστρατείες συλλογή υπογραφών. Η ΠΕΠ θα πρέπει να πω ότι είναι από το λιγότερο φιλικό για χρήση σύστημα που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ, γιατί ποτέ δεν, δεν είχε και στόχο να είναι αποκλειστικό. Νομίζω ότι η Περιτά αποκλείει τους ε, πολίτες εκτός ΕΕ και τους νέους. Επίσης, νομίζω ότι αποκλείει πολλούς πολίτες ΕΕ που ζουν εκτός ΕΕ και πολλούς Ιρλανδούς πολίτες οι οποίοι υποχρεώθηκαν να μεταναστεύσουν και έχουν ε, πάρα πολλούς λόγους να ασχολούνται με πολλά θέματα της πολιτικής ΕΕ. Εμείς θα παρακολουθήσουμε στενά το θέμα αυτό μετά την αξιολόγηση και υποστηρίζουμε το αίτημα για να θεώρηση του εργαλείου. Θα πρέπει λοιπόν να περιλάβουμε και την πρωτοβουλία εδώ για την ενιαία έδρα και να δούμε τα, και τα πολλά εκατομμύρια που πανούνται που κατασπαταλούνται για αυτό το περιοδεύοντα θεία. Σου ευχαριστώ. Έχουμε επισκέπτη σήμερα, λέει Πρόεδρο, και η συζήτηση αυτή του αφορά ιδιαίτερα, γιατί αυτή η πρωτοβουλία είναι στα δικά σας χέρια. Είναι ένα εργαλείο πολύ χρήσιμο και θα πρέπει να το χρησιμοποιήσετε. Ο κύριος Γιακολίνο έχει το λόγο τώρα, για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, είναι αλήθεια ότι μια Ευρώπη η οποία έχει ιδρυθεί στο δικαίωμα στα δικαιώματα των πολιτών χρειάζεται ένα εργαλείο όπως αυτό που δημιουργήθηκε, δηλαδή του δικαιώματος της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Ακούσαμε τους συναδέλφους μας και κυρία Μάλστρομ νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το εργαλείο αυτό καταγράφει κάποιες ε, δυσκολίες, κάποιες δυσκινησίες και δυσχέρειες. Είναι αλήθεια ότι κάποιες χώρες δεν συμμετείχαν με υπεύθυνο τρόπο στις εκστρατείες, ακόμα και στις ενημερωτικές. Υπάρχουν γραφειοκρατικές δυσκαμψίες και υπάρχουν δυσκολίες σε σχέση με το λογισμικό που χρησιμοποιείται, το οποίο προκάλεσε κάποιες δυσκολίες στην χρήση, έστω και αν ενδιάμεσα υπήρξε κάποια προσαρμογή του. Αν υπάρχει λοιπόν κάποια σκέψη που θα πρέπει να κάνουμε μετά από τις μέχρι τώρα παρεμβάσεις που ακούσαμε είναι το ότι επιβάλλεται μια τροποποίηση ενός ε, κανονισμού ο οποίος προωθεί περισσότερο την γραφειοκρατία παρά την ε, νέα πρωτοβουλία ή την γενοτόμα πρωτοβουλία των ε, πολιτών. Νομίζω ότι η ίδια η Κομισιόν θα έπρεπε να ενισχύσει τη δική της την δραστηριότητα μέσω συμβολής δική τη σε αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει επίση να ενθαρρύνουμε τι ε, χώρε μέλη και το Συμβούλιο θα έπρεπε να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία με μεγάλη όθηση, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Υπήρξαν βέβαια πρωτοβουλίε οι οποίε ε, στέφθηκαν με επιτυχία και ε, αναφέρθηκε το δικαίωμα για το νερό κλπ. Βασικά δικαιώματα και βασικές ελευθερίες θα μπορούσαν να ενισχυθούν περαιτέρω μέσω της προσφυγής της υπεύθυνη των πολιτών για θέματα όπως η ευημερία, ο πολιτισμός, η τοπικότητά τους θα μπορούσαν να προτείνουν σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες αν θα πρέπει λοιπόν να αναθεωρηθεί ο κανονισμός, αν θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια ατζέντα, ευρωπαϊκή ατζέντα για τους πολίτες, τότε οι πολίτες θα μπορούσαν πραγματικά να, οι ίδιοι να σχηματίσουν μια ευρωπαϊκή ατζέντα των προ, προτεραιοτήτων που οι ίδιοι θα ήθελαν να δουν να υλοποιούνται και που ενδεχομένως τα θεσμικά όργανα δεν ακολούθησαν μέσω των δραστηριοτήτων τους. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη ευελιξία. Τώρα ε, για την συλλογή των υπογραφών online, ακούσαμε διάφορες απόψεις. Οι πολίτες δεν θα πρέπει να αντικείμενο κοροϊδίας, δεν θα πρέπει να τους αρνούμαστε τα ίδια βασικά δικαιώματα και ελευθερίε που όπω προβλέπει και ο κανονισμό θα πρέπει να του παρέχονται. Ο κανονισμό ο οποίο θα πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να γίνει πιο ευέλικτο και πιο εύκαμπτο και ταυτόχρονα να παρέχει σημαντικέ και συγκεκριμένε δυνατότητε πρόσβαση σε πληροφορίε οι οποίε είναι απαραίτητε ώστε να γίνει το εργαλείο αυτό απτό και με προσθέμενη αξία. Αυτό θέλουμε λοιπόν. Μια Ευρώπη όπου οι πολίτες θα μπορούν να εκφέρουν την απόψή τους και ιδιαίτερα οι νέοι πολίτες. Να θυμίσω ότι συχνά έχουμε μεγάλη διαφορά μεταξύ και απόσταση μεταξύ των νέων πολιτών της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών οργάνων. Θα πρέπει λοιπόν οι νέοι να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που θα διαμορφώνει τις δραστηριότητες τους. Αυτό θα έχει τεράστια σημασία. Καταλήγω, Πρόεδρε, με μια έκκληση προς την κυρία Μάλστρομ, η οποία ανέκαθεν επέδειξε μεγάλη ευαισθησία και διαθεσιμότητα. Είμαι πεπισμένο ότι η Κομισιόν θα πρέπει να γίνει προωθητή αυτών των απαραίτητων πρωτοβουλειών που χρειαζόμαστε αφενό για να διασφαλίσουμε το γεγονό ότι οι χώρε μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν προ την κατεύθυνση αυτή και αφετέρου να απλουστεύσουμε με συγκεκριμένο και αυτό τρόπο ένα κανονισμό ο οποίο θα πρέπει να αποτελεί μια βασική πτυχή της συμμετοχής, της δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκυγιόμ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ. Και εγώ χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα απολογισμό ενδιάμεσο ε, της ε, πρωτοβουλίας Ευρωπαίων πολιτών, που είναι πάρα πολύ καινούριο βέβαια μέσα, όσο και σημαντικό. Ε, το είπατε και εσείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, συμμετείχε πάρα πολύ ενεργά ε, στην εκπόνηση του κανονισμού και ενδιαφέρεται να πετύχει το μέσο. Πολλοί όμως αναρωτήθηκαν για τα προβληματικά στοιχεία. Δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή αυτή η πρωτοβουλία, γιατί δεν την προωθούν και πολλοί τα κράτη-μέλη. Θα επανέλθω σε αυτό. Το σύστημα συλλογή υπογραφών είναι περίπλοκο. Υπάρχουν ζητήματα προστασία προσωπικών δεδομένων. Υπάρχουν ερωτήματα για τι προθεσμίε θεωρούνται σύντομες για να συλλεγούν οι απαραίτητες ε, υπογραφές. Ε, όλα αυτά φαίνονται φυσιολογικά ως απορίες και η διαδικασία μακροσκελεί στα μάτια των πολιτών. Βεβαίω θα πρέπει να υπάρχουν όλε οι ασφαλιστικέ δικλείδε για να μην υπάρχουν καταχρήσει και να προλαμβάνονται και να αποτρέπονται. Και τελικά μόνο οι πιο οργανωμένε ομάδε, τα λόμπι βασικά, που έχουν τη δυνατότητα να υπερβούν ορισμένα εμπόδια, καταφέρνουν να προωθούν τα ιδιαίτερα του συμφέροντα ει βάρος του συλλογικού συμφέροντος. Θα πρέπει λοιπόν κάθε πολίτη να μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία αυτή λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τούτων όλων λεχθέντων θα ήθελα να πω ότι Είμαι πεπισμένη ότι οι κυβερνήσει θα πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερε προσπάθειε για να κάνουν γνωστό αυτό το μέσο τη ΠΕΠ. Λυπούμε που δεν υπάρχει δήλωση του Συμβουλίου. Ελπίζω να μην είναι αυτό μήνυμα ε, του μικρού ενδιαφέροντος που δείχνουν ε, οι χώρες μέλη ε, για την πρωτοβουλία αυτή. Κυρία Ζαμπόσκα, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Όπως αναφέρατε και εσείς στην αρχή σας παρέμβαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει ε, την ε, περίοδο ε, για τις εννέα πρώτες πρωτοβουλίες πολιτών για να επιτρέψει την δραστηριοποίηση των πολιτών. Η 1η Νοεμβρίου είναι η νέα καταληκτική ημερομηνία, όπως είπατε. Όμως το Συμβούλιο των Υπουργών δεν δέχεται αυτή την ημερομηνία. Οι εθνικές κυβερνήσεις δεν γνωρίζουν πώς ακριβώς να θέσουν σε εφαρμογή την τροποποίηση τροποποίηση για την ημερομηνία. Πέραν αυτού δεν απαντούν σε μια κοινοβουλευτική ε, προφορική ερώτηση στα κατεπήγοντα και άρα μπορεί να ε, καταπέσουν εξαιτία τη τάση του Συμβουλίου κάποιε τέτοιε πρωτοβουλίε. Απευθύνομαι κυρίω σήμερα στο Συμβούλιο της Ένωση ζητώντα ε, άμεση απάντηση στην προφορική ερώτηση που έθεσα το 1905 του 2013 υποχρεούται το Συμβούλιο σε περίοδο τριών εβδομάδων να δώσει απάντηση σε δύο προφορικές ερωτήσεις. Αν δεν αποφανθεί για την νέα καταληκτική ημερομηνία για τη συλλογή υπογραφών για τις εννέα πρώτες πρωτοβουλίες, ε, θα σημάνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αρνείται να αποφανθεί και αυτό θα μας οδηγεί σε μεγάλη νομική ανασφάλεια εις βάρος ε, του εργαλείου της πρωτοβουλίας των πολιτών ε, επίτροπε. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο ε, κατόμπι συνεννόησης να δράσουν, τόσο ώστε να μην υπάρξει αυτή η νομική ανασφάλεια για τις εννέα ε, αυτές πρώτες πρωτοβουλίες και να μην υπάρξει νομικό κόλλημα. Ε, πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Κύριος Μάρτιν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, όπως και άλλοι βουλευτές Πιστεύω ότι η πρωτοβουλία των πολιτών έχει προοπτική να δημιουργήσει ένα δημόσιο χώρο όπου τα θεσμικά όργανα και οι πολίτε θα είναι σε διαρκή διάλογο. Επίση, οι πολίτε πολλών κρατών θα μπορέσουν διασυνοριακά να υπερασπιστούν τα συμφέροντά του και αντίθετα με τον κύριο Μπάτεν πιστεύω ότι υπάρχει ένα Δήμο Ευρωπαϊκό και αυτή η πρωτοβουλία τον ενισχύει. Νομίζω ότι βλέπουμε μια ξεκάθαρη δέσμευση σε σχέση με την πρωτοβουλία ε, των πολιτών και ξέρουμε ότι η Επίτροπο έχει αναλάβει προσωπική δέσμευση. Α συνεχίσει λοιπόν, να συνεχίσει να ασκεί πίεση, ούτω ώστε να απλουστεύσουμε και να βελτιώνουμε τη διαθέσιμη τεχνολογία. Επίση, να έχουμε μια κεντρική επιγραμμική ή σε απευθεία σύνδεση πλατφόρμα για τη συλλογή των υπογραφών. Ε, αναφερθήκατε και στο πρόβλημα του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Ιρλανδία. Ελπίζουμε αυτέ οι κυβερνήσει ε, να μειώσουν ε, το κατόφλι ε, για να μπορέσουν και οι πολίτες πολίτες ε, εκτός των δύο χωρών ε, να μετάσχουν στην πρωτοβουλία. Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνουν περισσότερα για την ενημέρωση των πολιτών από πλευράς Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα όπου υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Σινίζη νομίζω απουσιάζει και άρα η κυρία Εστρέλα για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συνθήκη της Λισαβόνας ενίσχυσε την συμμετοχική δημοκρατία και την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας είναι ένα θετικότατο εργαλείο, όπως ακούσαμε. Χρειάζεται απλούστευση των κανόνων και των διαδικασιών ε, που δυσχεραίνουν την υλοποίηση ε, του νέου αυτού θεσμού. Ε, επικροτούμε τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διευκόλυνση μιας εγνήσιας δημοκρατικής των πολιτών πολιτών στη διαδικασία λήψη αποφάσεων για, την ευρωπαϊκή, για τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Το ευρωπαϊκό έτος των πολιτών και σε αυτή την περίοδο όπου η Ευρώπη διέρχεται μια περίοδο βαθύτατης οικονομικής κρίσης αλλά και πολιτικής κρίσης και κρίσης αξιών είναι απαραίτητο να εμβαθύνουμε το διάλογο ανάμεσα στους ε, ε, ε, ε, τάγους και τους πολίτες έτσι δημιουργούμε ένα νέο δρόμο για την Ευρώπη που απηχεί και τις προσδοκίες των πολιτών που, έτσι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη και στα επιμέρους κράτη-μέλη έχουν ε, απογοητεύσει τους πολίτες ε, και βλέπουμε ε, ότι διαδηλώνουν στους δρόμους πολίτες για να ακουστεί η φωνή τους. Ας χρησιμοποιήσουμε το νέο εργαλείο. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Κλέβα Κέκους τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η δυνατότητα στενότερης συνεργασίας, η δυνατότητα συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών στη συζήτηση για θέματα που αφορούν την καθημερινότητά τους και ε, μάλιστα πάρα πολύ σοβαρά είναι σημαντικότατη. Θα πρέπει να φτάνουμε σε όλους τους πολίτες και σε εκείνους κυρίως που δεν συμμετέχουν συνήθως στα κοινά, δεν συμμετέχουν στις αποφάσεις για τα ευρωπαϊκά θέματα. Ακριβώς λοιπόν με την ε, πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών σε αυτούς τους πολίτες απευθυνόμαστε και σε αυτούς τους πολίτες φτάνουμε. Θα πρέπει τώρα όμως να ε, τους δίνουμε ένα εργαλείο πιο προσωπικό, πιο πρακτικό για να μπορούν να συμμετέχουν και να επιθυμούν και να συμμετέχουν. Υπάρχουν πολλά τεχνικά που πρέπει να βελτιωθούν. Το σύνολο σύστημα γενικότερα, 30 πρωτοβουλίες τρέχουν αυτό το καιρό και μόνο μία έχει ήδη συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο υπογραφές. Αυτό σημαίνει ότι κάτι χωλαίνει στο σύστημα. Αλλά βέβαια τώρα μόνο 12 μήνες λειτουργίας έχει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοφεράτη παρακαλώ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, όταν αποφασίστηκε στη Λισαβόνα να θεσπιστεί το εργαλείο αυτό της ΠΕΠ είχαμε κάνει επιδείξη μεγάλης διορατικότητας γιατί έχουμε ένα εργαλείο το οποίο έχει παρουσιάσει ένα τεράστιο δυναμικό και προσεγγίζει τους πολίτες και συγνώριζεται πολύ καλά πόσο το χρειαζόμαστε αυτό σε αυτή την φάση οικονομικής κρίσης όπου τα κοινωνικά προβλήματα κάνουν πολλούς πολίτες να υποφέρουν οι οποίοι βλέπουν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εχθρότητα όργανα τα οποία δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα αιτήματά τους. Ενώπιν λοιπόν αυτού του δυναμικού που έχει αυτό το εργαλείο, δεν θα πρέπει όμω να αποκρύπτουμε του περιορισμού του και εσεί αναφερθήκατε σε αυτού. Οπότε θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα άμεσα. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί η αναθεώρηση για το 2015 του εργαλείου. Θα πρέπει να γίνει νωρίτερα. Είναι προφανέ ότι είναι ελάχιστα γνωστό αυτό το εργαλείο και είναι παράδοξο ότι ένα μεγάλο εργαλείο άμεση δημοκρατία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλήρω επειδή οι πολίτε δεν γνωρίζουν την ύπαρξή του και ακόμα λιγότερο αγνοούν την πραγματική του λειτουργία. Και τέλος θα πρέπει οι πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν προωθηθεί να γίνουν και αυτές ε, νομοσχέδια γιατί εάν οι πολίτες οι οποίοι συμμετέχουν σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι ακόμα τέλεια όσον αφορά ε, το θέμα της αναγνώρισης του εργαλείου για να υποδείξουν στα θεσμικά όργανα χρόνους, διαδικασίες κτλ. και αυτά δεν ρυθμίζονται, δεν ε, λύνονται, τότε θα έχουν εχθρική στάση προς το εργαλείο. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό νομίζω σύντομα να μετατραπούν κάποιες από αυτές τις πρωτοβουλίες που έχουν κατατεθεί σε νομοσχέδια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στη δικασία Δίνω το λόγο στον κυριο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Στα όσα υπόθηκαν να προσθέσω κι εγώ μετά από την περιήγηση την αναλυτική που έκανα και στον επίσημο διαδικτυακό χώρο, το Μητρό που έχει φτιάξει η Επιτροπή για αυτή την πρωτοβουλία, το οποίο παρεμπιπτόντως είναι πολύ χρηστικό και θέλω να συγχαρώ την Επιτροπή γι' αυτό ότι εκεί μπορεί κανεί να δει πολύ καλέ πρωτοβουλίε και πολύ καλέ ιδέε. Δεν είναι πράγματι πολλέ, είναι όμω σημαντικέ και δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε θέλουν να πάρουν την Ευρώπη στα χέρια του και οι προτάσεις αυτές, αν τις μελετήσει κανείς, είναι περισσότερο προωθημένες και πρωτοποριακές πολλές φορές και από εκείνες τη Επιτροπής και των κρατών μελών. αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε αισιόδοξοι. παρότι οι προτάσει δεν είναι πολλές, βλέπει κανείς ότι μετά την συνθήκη της Λισαβόνας που καθιερώνει πλέον την αρχή της λογοδοσίας, την κρίσιμη αυτή περίοδο που αμφισβητούνται σε κοινωνικό οικονομικό πολιτικό επίπεδο τα πάντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή η προσπάθεια μπορεί να αποδώσει καρπούς. βεβαίως δεν είναι αρκετό μόνο να την τονίσουμε επικοινωνιακά έχει πολύ μεγάλη σημασία όπως υπόθηκε και από τον κύριο κοφεράτη προηγουμένως να υιοθετηθούν κάποιες από αυτές τις προτάσεις να μπορέσουμε να δείξουμε εν της πράγμαση ότι δίνουμε λόγο στους ευρωπαίους πολίτες. έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε ας είμαστε όμως σας ευχαριστώ. Ε, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, θα είναι συνάρτηση της έκβαση των προσπαθειών για την κατάργηση του δημοκρατικού ελλείμματο. Χρειαζόμαστε συστηματικές, συστημικές συγγνώμη, λύσεις για να ενισχύσουμε το δημόσιο χώρο διαλόγου, αυξάνοντας τη συμμετοχική διάσταση της δημοκρατίας. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, διαθέτει αυτό το θεσμό, αλλά δεν είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία. Συλλέγονται οι υπογραφές ε, για ε, το ελάχιστο εισόδημα παραδείγματος χάρη. Είναι δημαγωγικού χαρακτήρα. Δηλαδή όλοι οι πολίτες ε, θα λαμβάνουν 500 ή 600 ευρώ από το κράτος ανεξαρτήτως οικονομικών πόρων. τι, ε, νομίζουν ότι τα κράτη τυπώνουν ε, συνέχεια χρήματα, δεν παράγονται. Ε, θα δημιουργηθεί μια τεράστια τρύπη, τρύπα στην κοινωνία. Όταν θα λάβετε αυτή την πρωτοβουλία, Επίτροπε, πώς θα αντιδράσετε. Ευχαριστούμε, κυρία Τούρμου, για ένα λεπτό żeby inicjatywa obywatelska była naprawdę instrumentem dla Ευχαριστώ. Εγώ επιθυμώ η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών να είναι ένα εργαλείο στα χέρια των πολιτών που μπορούν να συμμετέχουν βέβαια οι εκλογές, αλλά μέχρι στιγμής το μόνο εργαλείο που έχουν είναι αυτό. Δεν είναι για τους πολιτικούς φτιαγμένη η πρωτοβουλία. Εμείς έχουμε νομοθετική δραστηριότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Είμαστε νομοθέτες. Ε, ανησυχώ που ακούω διάφορε φωνές εδώ βουλευτών οι οποίοι ζητούν να περιορίσουμε αυτό το εργαλείο. Να μην έχουν, λέει, την ευκαιρία να συμμετέχουν πάρα πολύ τα συνδικάτα ή τα λόμπι, οι ομάδες πίεσης. Μα κυρία Επίτροπε, θα πρέπει να το αφήσουμε αυτό το μέσο στα χέρια των πολιτών και όχι σε ε, οργανωμένες ομάδες συμφερόντων. Μήπως να ξανασκεφτούμε τον προσανατολισμό της πρωτοβουλίας αυτής. Να φροντίσουμε όλοι να ενημερώνουμε τους πολίτες. Είναι καταπληκτική αυτή η δυνατότητα. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάντενμπαχ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Πίτροπε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την άμεση και ενεργή συμμετοχή των πολιτών ε, σε αυτή ε, την πρωτοβουλία. Τώρα είναι ακόμα στα σπάργανα, εξού και οι παιδικές αρρώστιες που συνοδεύουν την κατάσταση αυτή. Ε, ακριβώς όμως μετά τη συζήτηση θα πρέπει να δούμε συνολικά την κατάσταση. Χαίρομαι που βλέπω και ομάδες επισκεπτών εδώ. Το πρόβλημα δεν είναι βέβαια δικό τους άμεσα, αλλά θα πρέπει να εξηγούμε και στο Κοινοβούλιο και να αυξάνεται η δυνατότητα ε, περισσότερων επισκεπτών στο Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα για μαθητές. Βέβαια δεν φταίτε εσείς κυρία Πρόεδρε, αλλά το λέγω. Το παρλαμεντάριο μου στις Βρυξέλλες έχει δωρεάν είσοδο ελεύθερη και θα ήθελα να γίνει γνωστό αυτό και επίση η δυνατότητα συμμετοχή σε δημόσιε ακροασει μαζί με του πολίτε, μαζί με τι πρωτοβουλίε των πολιτών. Όλα αυτά θα πρέπει να τα διαδώσουμε, να τα διαφημίσουμε διότι ε, δεν χρησιμοποιούνται παρκώ ακόμα πρέπει να σας πω ότι η καθημερινότητα των βουλευτών εδώ μας υποχρεώνει να έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο για να φερώνουμε στους πολίτες μας και αυτό να το σκεφτούμε. Εγώ θεωρώ ότι εκπροσωπώ τους ψηφοφόρους μου, άνδρες και γυναίκες και τους Ευρωπαίους πολίτες συνολικότερα. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Λούχαν τελευταίος, για 1,5 λεπτό. Ναι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, μετά από ένα χρόνο λοιπόν ε, πρωτοβουλίας Ευρωπαίων πολιτών βλέπουμε ότι έχουν συλλεγεί υπογραφές μόνο για μία πρωτοβουλία όσες χρειάζονται. Ε, είναι πάρα πολύ περίπλοκη λοιπόν η ε, διαδικασία και ούτε λόγος γίνεται για εναρμόνιση σε επίπεδο κρατών μελών. Οι πολίτες αισθάνονται αποκλεισμένοι από τη χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής. Χρειάζεται οπωσδήποτε εναρμόνιση των κριτήριων και των διαδικασιών σε επίπεδο κρατών μελών. Επίσης θα πρέπει να βρούμε μια πλατφόρμα, ένα λογισμικό που να είναι πιο φτηνό και πιο εύκολο στη χρήση και εδώ να λάβουμε υπόψη τη δυνατότητα το σύστημα να το ε, οργανώσουμε κεντρικά ε, με κύριο υπεύθυνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης να υπάρχουν σημεία επαφής για ενημέρωση, για πληροφόρηση των πολιτών για ε, διάφορα επιμέρους γραφεία. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται εδώ το Καζιά και το λόγο έχει η Επίτροπος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Να κυρίε και κύριοι, για αυτή τη θαυμάσια συζήτηση. Νομίζω ότι είπε, πολύ συμφωνούμε ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την ενίσχυση τη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και να κάνουμε του πολίτε μετέχοντε και συμμετόχου στη λήψη αποφάσεων για σημαντικά θέματα που του απασχολούν όπου και να ζουν στην Ένωση. Και ελπίζω σύντομα μία από αυτέ τι πρωτοβουλίε θα κατατεθεί στην Κομισιόν ώστε να αρχίσουμε να την προωθούμε. Αυτό αποτελεί μια επιτυχία βέβαια, αλλά όπω εσεί ε, αναφέρατε και όπω είπα και εγώ στα σχολιά μου, υπάρχουν κάποιε παιδικέ ασθένειε. Κάποιε από αυτέ αφορούν κάποια αρχικά προβλήματα και θα πρέπει να τα εξετάσουμε. Βεβαίω έχουμε ευθύνη στην Κομισιόν εμεί για την πρόθεση τη ε, πρόταση και Εσεί και το Συμβούλιο ως ε, συνομοθέτε για την υπόλοιπη δουλειά. Εμεί ήδη έχουμε αποφασίσει να ε, συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε το σύστημα συλλογή υπογραφών online, λύση η οποία δεν είναι οριστική και ιδανική, αλλά αυτό γίνεται μέχρι να βρούμε μια τελική λύση. Και θα πρέπει να δούμε επίση κατά πόσο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα κεντρικό ή κεντρικοποιημένο σύστημα, κάτι το οποίο ανέφεραν πάρα πολύ στα σχολεία του εδώ και θα πρέπει να το εξετάσουμε. Η Κομισιόν συμφωνεί επίση απόλυτα και έχει ζητήσει από τις χώρες ε, μέλη να το κάνουν ότι θα πρέπει να μειωθούν τα κατόφλια, ε, τα αριθμητικά για την συλλογή των υπογραφών. Είμαστε επίσης σε επαφές με τις χώρες ε, μέλη για την επέκταση των προθεσμιών που αναφέραν κάποιοι από εσά και είχαμε επικοδομητικό διάλογο για αυτό το θέμα και είμαι πεπισμένη ότι θα βρούμε και επ' αυτού μια λύση πολύ σύντομα. Ο κ. Σέμα είπε, μάλλον με ρώτησε κάτι σε σχέση με την πρωτοβουλία στην οποία συμμετείχα εγώ οι απόψεις μου είναι ξεκάθαρες νομίζω και γνωστές για αυτό το θέμα. Η σωστή λοιπόν απάντηση στο ερώτημά σας είναι ότι οι αλλαγές στη συνθήκη δεν περιλαμβάνονται στα, στο πεδίο των προτάσεων. Αυτή είναι η χρονιά των πολιτών. Κατά κάποιο τρόπο κάθε χρονιά θα πρέπει να είναι η χρονιά των πολιτών αλλά σε αυτή ακριβώς τη χρονιά των πολιτών θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάποια πράγματα σοβαρά. Εμείς από την Κομισιόν, η, η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ και άλλοι, και εγώ και άλλοι συνάδελφοι, ενεργά επισκεφτόμαστε χώρες μέλη, επισκεπτόμενοι σχολεία, οργανώσεις, ε, ε, ώστε να προωθήσουμε αυτή την πρωτοβουλία και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε αυτό, επειδή πραγματικά αποτελεί μια θαυμάσια πρωτοβουλία. Εσείς ως η ερετή του ευρωπαϊκού λαού έχετε και τη δική σας ευθύνη ώστε να το προωθείτε με κάθε ευκαιρία και όχι μόνο σε τακτική βάση, αλλά και ενώπιση των ευρωπαϊκών εκλογών που αποτελούν μια θαυμάσια ευκαιρία γι' αυτό. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να βελτιώσουμε τη λειτουργία αυτή τη πρωτοβουλία, να την διαδώσουμε, γιατί αποτελεί ένα πολύ ισχυρό και θαυμάσιο εργαλείο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ε, συζήτηση. Είμαι βέβαιος ότι θα μεταφερθούν όλες οι παρεμβάσεις στον Αντιπρόεδρο Σεύκοβιτς και θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα αυτό στην Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ελπίζω οι επισκέπτες να κατάλαβαν όλοι ότι περιμένουμε αν θέλουν να καταθέσουν πρωτοβουλίες ε, σε συνεργασία με πολίτες 7 χωρών. Ε, Μην διστάσετε λοιπόν, ε, περιμένουμε